Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take... Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Τότε θα κάνουμε ξαναδιαβά... Ξανα... Όλο και περισσότερο θόρυβο κάνουμε εδώ.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 και από του διερμηνείς σα να σα ενημερώσουμε ότι βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων λόγω τη εργασιακή διανέξης με τη διοίκηση για τι συνθήκες εργασία μα. Σε κάποιε καμπίνες έχουν επιστατευτεί όλοι οι διερμηνείς και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν. Αυτό ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμά μα στην απεργία και συνιστά διάκριση προ τι υπόλοιπε γλώσσε. Ω εκ τούτου, η ελληνική καμπίνα δεν θα προχωρήσει στη στάση εργασία για τη σημερινή συνεδρίαση σε ένδειξη ελληνική. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Βον πριν την ψηφοφορία ευχαριστεί τη γραμματεία και όλου του κοιόδη. Ε, που είπαν ότι είναι καλή η έκθεση θα γνωρίζετε από τη συζητήση μας στην Επιτροπή και τη στήριξη της, ε, ότι θα στείλουμε μια Επιτροπή ε, Αναζήτησης ε, Στοιχείων και νομίζω πως αυτό ε, γίνεται σε μια πολύ κατάλληλη στιγμή γιατί μέσα από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προτείνουν να στηριχτεί η χρηματοδότηση για τη διαδικασία ειρήνευσης στη Βόρεια Ιρλανδία. Σήμερα έχουμε καμιά καλή ευκαιρία να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι επίσης πιστεύουμε πως αυτό το πρόγραμμα είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί και μετά το 2020 και ελπίζω πως σήμερα θα έχουμε θετική ψηφοφορία από τους συναδέλφους και αν είναι δυνατόν και ομόφωνη ψήφο, ώστε να στείλουμε ισχυρό μήνυμα προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ψηφίσουμε. Και ξεκινάμε με την τροπολογία υπαριθμών 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε να ελέγξουμε την τροπολογία 1. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. First of Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Okay. We, we continue now with the amendment. Συνεχίζουμε με την τροπολογία υπαριθμών 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 με προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά της προφορικής, όχι. Οπότε ψηφίζουμε την 15 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοντ 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ε, τροπολογία 41 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 41 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Και απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Τέλος. Και εγκρίνεται η έκθεση λοιπόν. χαρτίρια κύριε Βόν. Επόμενη έκθεση είναι αυτή που είναι του συναδέλφου Πασκαλαρίμό, ειδικά μέτρα για την Ελλάδα. Κύριε Αριμό, θέλετε κάτι να πείτε πριν την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ πως η έκθεση αυτή είναι ένα δείγμα της αλληλεγγύης της Ευρώπης, είναι ένα, είναι κάτι που αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής και απόδειξη του ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει ε, συνένεση και συνεργασία σε όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για αυτή την έκθεση, να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για την εξαιρετική συνεργασία, καθώς και τους δικούς μου συνεργάτες. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ. Α ξεκινήσουμε τώρα την ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Α, συγγνώμη. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Με προφορική τροπολογία. Υπάρχει ένσταση για την προφορική. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν μαζί με την προφορική για την 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 είναι ταυτόσιμη με το 16. Πάμε λοιπόν στην 18. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Να ελέγξουμε τη 19. Ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται.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 56 καταπίπτη, Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τελείωσε λοιπόν και η ψηφοφορία για σήμερα. Και συνεχίζουμε. With με την ανταλλαγή απόψεων. Αρχικά είχαμε ζητήσει να γίνει μια ακρόαση, όμως νομίζω πως ε, αν δεν κανείς τον κατάλογο των ε, ομιλητών και των παρουσιάσεων είναι σχεδόν σαν να κάνουμε ακρόαση. Οι συγητές ζήτησαν ε, αυτήν την ανταλλαγή απόψεων και η πλειοψηφία των μελών ε, της Επιτροπής μας επίσης. Θα γίνει λοιπόν ανταλλαγή απόψεων για μια νομοθετική πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού ε, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το αποθεματικό απόδοσης. Έχει πολύ μεγάλο τίτλο το θέμα, οπότε λοιπόν σας έκανα έτσι μια σύντομη παρουσίαση. Η πρόταση αυτή στόχο έχει να μεταρρυθμίσει τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων έτσι ώστε να επιδέψει την ύπαρξη αποθεματικού επιδόσεων να χρησιμοποιηθεί για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για συγκεκριμένες προτεραιότητες που θα τεθούν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Η πρόταση αναφέρεται ιδιαίτερα στο άρθρο 22.1α, 22.8 και 23α του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, όπου τίθενται οι αρχές χρήσης του ε, Ταμείου Συνοχής για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι διατάξεις του κανονισμού κοινών διατάξεων αφορούν τους ορισμούς, την χρέωση υποβολής ε, εκθέσεων μεταξύ άλλων και κατόπιν ε, πρότασης των συντονιστών έχουμε καλέσει αρκετού εμπειρογνώμονε για να γίνει ανταλλαγή απόψεων πάνω στι διαφορετικέ πτυχέ του θέματο αυτού. Υπάρχει ειδική ημερήσια διάταξη για το θέμα αυτό. Θα ήθελα Καταρχάς, να δώσω το λόγο στον κύριο Φονμπρέσκα. Έχουμε καιρό να σας δούμε. Σας δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο για να μας εξηγήσετε με δύο λόγια την πρόταση της Επιτροπής. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πάρω ξανά το λόγο και σας υπόσχομαι αυτή τη φορά να είμαι πιο σύντομος από το πρωί. Με μεγάλη μου χαρά έχω τη συνάδελφο Μέρι Μακάρθη, η οποία είναι από την Υπηρεσία στήριξη Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων τη ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία νομίζω θα μας δώσει επιπλέον πληροφορίες για πτυχέ των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ε, που αναφέρονται στην πρόταση αυτή. Όπως και σήμερα το πρωί έχω και τώρα διαφάνειες, θα σας ε, Κάθε λοιπόν, θα σας κάνω μια συνοπτική παρουσίαση των διαφανειών αυτών και θα αρχίσω λέγοντα, εξηγώντας γιατί έχει γίνει αυτή η πρόταση. Καταρχάς, οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Και τι εννοώ με αυτό. Για παράδειγμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δυσκολία στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Πολλές φορές δραστηριοποιούνται σε δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον ή δυσκολεύονται ε, να ε, στήσουν τις επιχειρήσεις τους, ε, να γίνονται καθυστερήσεις στις δικαστικές αποφάσεις και ακόμα και αν ε, στηρίζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ευρωπαϊκές επενδύσεις, πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο του έργου τους. Αυτό λοιπόν συνιστά την ανάγκη για διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις και γι' αυτό Έχουμε αυτή τη στιγμή την πρόταση της Επιτροπής η οποία επιτρέπει την ύπαρξη ενός μηχανισμού που θα παρέχει κίνητρα για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις χρησιμοποιώντας ε, αντίστοιχα κονδύλια. Θα ήθελα καταρχάς να σας ε, πω ότι αυτό είναι κάτι προαιρετικό όπως βλέπετε. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει το μέσο αυτό. Είναι λοιπόν ε, κάτι που έχει προαιρετικό χαρακτήρα. Μπορούν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν προαιρετικά το αποθεματικό αυτό για να ε, δρομολογήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Το δεύτερο που ήθελα να τονίσω, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της διαφάνειας, είναι ότι δεν τίθεται υποαμφισβήτηση ε, ο προσανατολισμός των επιδόσεων αυτών. Το αποθεματικό αυτό διατηρείται για τα προγράμματα τα οποία ήδη υπάρχουν, ήδη τρέχουν, δεν γίνονται κάποιες αλλαγές εδώ, θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ισχύ, δεν αμφισβητείται λοιπόν τίποτα. Τώρα, πώς λειτουργεί το μέσο αυτό. Σύμφωνα με την πρότασή μας, όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει, να βρω και που είμαι. Νομίζω έτρεξα λίγο. Α, εδώ είμαι. Όταν λοιπόν ένα κράτος μέλος θέλει να το χρησιμοποιήσει, πρέπει να υποβάλει μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, αναθέσει ένα μέρος ή όλο το αποθεματικό για μια συγκεκριμένη ανάληψη υποχρεώσεων. Θα αναφέρονται τα συγκεκριμένα μέτρα που θέλει να υλοποιήσει, οι στόχοι, που ε, πρέπει να επιτευχθούν και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα εδώ έχει ένα σημαντικό στοιχείο. Ε, υπάρχει ένα ανώτατο όριο τριών ετών. Γιατί τρία χρόνια. Διότι πρόκειται για πιλωτικό πρόγραμμα δεν θέλουμε λοιπόν να περιπλέξουμε τα πράγματα και να ε, προσπαθήσουμε να κάνουμε το κατόρθωτο. Εστιάζουμε κυρίως σε ε, βραχυπρόθεσμα προγράμματα για να δημιουργήσουμε ε, ένα προηγούμενο, να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το εργαλείο πριν το 2020. Όταν ένα κράτος μέλος λοιπόν επιλέγει να το χρησιμοποιήσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει την πρόταση. Μετά από διάλογο με τα κρατημέλη, υπάρχει εκτελεστική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζονται τα ε, καταβληθέντα ποσά και ε, υλοποιούνται πλήρως τα προγράμματα. Και προς αποφυγή περαιτέρω γραφειοκρατίας υπάρχει έλεγχος, υπάγεται πλήρως τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη υποβάλλουν εκθέσεις μέσω των εθνικών προγραμματών μεταρρύθμισης σε εμάς κάθε χρόνο. Αναφέρονται ε, τα ορόσημα, οι στόχοι και κατόπιν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ε, παράσχει στήριξη στους ε, τομείς όπου τη ζητείτε. Όπως σας είπα, τα κράτη-μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια της επιλογής και αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι φυσικά το, δεν αποφασίζει το κράτος μέλος, διότι τα κονδύλια αυτά πρέπει να ε, βγουν από κάποιο πρόγραμμα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι και οι περιφέρειες που θα αναλάβουν αυτά τα προγραμματά και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να εγκρίνουν την πρόταση αυτή προτού γίνει οτιδήποτε. Όλοι λοιπόν οι εταίροι σε όλα τα επίπεδα συμπεριλαμβάνονται στην διαδικασία προτού αντιληθούν κονδύλια από κάποιο πρόγραμμα συνοχής. Τον τελικό λόγο λοιπόν έχουν ε, όσοι έχουν και τα κονδύλια. Το πιο σημαντικό είναι το τελευταίο σημείο στη διαφάνεια που βλέπετε. Θέλουμε άμεση διαχείριση για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Και γιατί. Διότι θεωρούμε πως ε, διαφορετικά θα γίνει πολύ δύσκολο, χρονοβόρο ε, και περίπλοκο το να εφαρμόσουμε όλο το πρόγραμμα και να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις ε, για την υλοποίηση των πιλωτικών αυτών προγραμμάτων. Να πω δύο λόγια για τις μεταρρυθμίσεις τώρα, αν και είμαι σίγουρος ότι η Μέρη θα σας ε, πει περισσότερα. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουν αποτέλεσμα το οποίο θα αναφέρεται στους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Χρειάζονται φυσικά ε, κίνητρα, όμως ε, δεν υπάρχει εδώ κάποια δυνατότητα άμεσης αποζημίωσης για το κόστος μεταρρυθμίσεων. Όπως σας είπα, το μόνο που γίνεται εδώ είναι να παρέχονται κίνητρα. Αυτή τη λογική ακολουθούμε και γι' αυτό θα υπάρχει μία ενιαία ενίσχυση όταν ε, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Πότε θα γίνει όλο αυτό. Σύμφωνα με την πρότασή μας, αυτό θα συμβεί στο πλαίσιο του επόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δηλαδή, ελπίζουμε τα κράτη-μέλη να μας ενημερώσουν στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων του 2019 για το αν προτίθενται ή όχι να χρησιμοποιήσουν το μέσο αυτό. Και αυτό διότι φυσικά η διαδικασία αυτή συνεπάγεται κάποιες τροποποιήσεις, πρέπει να βγουν κονδύλια από άλλα προγράμματα, να γίνουν αναλήψεις υποχρεώσεων και φυσικά πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ε, του αποθεματικού επιδόσεων. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο της επόμενης χρονιάς, γιατί τότε θα ε, πιστωθούν ε, οι πόροι από το αποθεματικό. Μετά θα είναι πάρα πολύ αργά για να γίνουν αλλαγές ή τροποποιήσεις. Αυτά λοιπόν ως προς το χρονοδιάγραμμα και τις ε, προθεσμίες, νομικές προθεσμίες για τις ενδεχόμενες μεταφορές πόρων. Τώρα, για λόγους απλούστευσης. Δεν ε, επιδέχεται το πρόγραμμα αλλαγές. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα ποσά και αυτό φυσικά σημαίνει ότι οι στόχοι πρέπει να είναι φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστικοί. Ελπίζουμε επίσης να ληφθούν υπόψη και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες στο πλαίσιο της απόφασης. Και ορισμένα τελικά σχόλια. Επιτρέψτε μου. Τι σημαίνει αυτό για τις πληρωμές. Δεν υπάρχει λοιπόν αποζημίωση δαπανών, γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχουν και κανόνες επιλεξιμότητας. Δεν επιστρέφονται λοιπόν χρήματα από δαπάνες, δεν υπάρχει ανάγκη συγχρηματοδότησης. Υπάρχει επίσης, δεν υπάρχει επίσης προχρηματοδότηση ούτε και ε, καταβολές για μερική υλοποίηση. Θέλουμε λοιπόν, όπως σας είπα, να είμαστε όσο το δυνατόν απλούστεροι. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ανάγκη για διάφορες πρόσθετες λειτουργίες, ελέγχους, επαληθεύσεις. Η μόνη επαλήθευση που πρέπει να γίνει είναι μια αξιολόγηση για το αν έχει υλοποιηθεί ε, κάποια ανάληψη υποχρεώσεων, ε, αν έχουν, γίνει οι μεταρρυθμίσεις. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι στην ουσία η προσέγγιση μας είναι απλή, είναι ε, ερώτηση που επιδέχεται ένα ναι ή ένα όχι ως απάντηση. Η τελική απόφαση βέβαια εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως υπάρχει και η δυνατότητα το κράτος μέλος να υποβάλει μια πρόταση, να επιχειρηματολογήσει γιατί ας πούμε θέλει, ε, γιατί θέλει να υλοποιήσει μια μεταρρύθμιση, γιατί και το αν η μεταρρύθμιση έχει ή όχι υλοποιηθεί. Τέλος. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι. Δεν γίνεται να μεταφερθούν οι πόροι πίσω στα προγράμματα αυτά, διότι θα έχουν ήδη αποδεσμευτεί. Αυτά λοιπόν, νομίζω πως θα σταματήσω εδώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιορτανόβα, υπεύθυνη για την μακροπεριφερειακή στρατηγική από την μόνιμη αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας παρουσιάσει μια δήλωση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που, για την πρόσκληση που απευθύνατε προς ε, το Συμβούλιο στη σημερινή συνεδρίαση. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση ε, για την πρόοδο που έχει σημειωθεί ε, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο θεωρεί πολύ σημαντική την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα των ερευνητικών τομέων, ταμείων. Ε, είναι μεγάλη η πολιτική ε, σημασία και η λεπτότητα και η συνθετότητα αυτής της διαδικασίας στο πλαίσιο και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Παραμένει σημαντικό για το Συμβούλιο οποιαδήποτε μέτρα στον τομέα της ε, πολιτικής συνοχής να αφορούν την ε, προαγωγή ε, της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Η ομάδα εργασίας άρχισε να εξετάζει τον φάκελο στις 20 Φεβρουαρίου. Η πρώτη αντίδραση των, κράτη, κρατών μελών ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική με πολλά ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια είχαμε δύο συνεδριάσεις με γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 19 Μαρτίου ε, και 24 Απριλίου. Πέραν των γραπτών εξηγήσεων, και των συζητήσεων στην ομάδα εργασία, η πλειονότητα των κρατών μελών διάκειται αρνητικά ε, στην ε, πρόταση σε πολλά σημεία για το χρονοδιάγραμμα, μεταφορά ε, ποσών από το αποθεματικό επιδόσεων, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των πραγματεύσεων και η λεγόμενη δέσμευση μεταρρυθμίσεων. Βάσει των επιφυλάξεων των αντιπροσωπιών, αποφασίστηκε ο φάκελο να μπει στον πάγο μέχρι νεοτέρας και έτσι να δώσουμε τη δυνατότητα και στα κράτη-μέλη να λάβουν σε υπόψη την πρόταση για το επερχόμενο P-ΔΑΛΤΑ-ΠΗ και την κλαδική νομοθεσία για την πολιτική συνοχή. Δεν αναμένεται κάτι καινούριο υπό τη Βουλγαρική Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η δήλωση του Συμβουλίου, εξαιρετικά σαφής σύντομη και σαφής. Uh, Τώρα συνεχίζουμε με την κυρία Μέρι Μακάρθη που είναι διευθύντρια της μονάδας ε, στήριξης για τις Διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό να σας δείξω και τις ε, διαφάνειες. Έχω λοιπόν ετοιμάσει μια παρουσίαση με πολλές διαφάνειες, δεν θα σας τις ε, αναλύσω όλες, μην ανησυχείτε. Θα εστιάσω σε λίγες από αυτές τις ε, διαφάνειες για να τονίσω κάποια πράγματα. Καταρχάς λοιπόν θα μιλήσω για το ρόλο της υπηρεσίας στήριξης θετικών μεταρρυθμίσεων και το σχετικό πρόγραμμα. Μετά θα μιλήσω για θέματα όπως η διαφορά ανάμεσα στο πρόγραμμα και το εργαλείο επίτευξης των μεταρρυθμίσεων καθώς και τι γίνεται υπό τη στροποποίηση του CPR. Με συγχωρείτε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, λέει η Πρόεδρος. Όχι, ωραία λοιπόν. Έχουμε και την παρουσίασή σας και εμείς. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Και συνεχίζω. Θα περάσω αμέσως σε αυτή την εδώ τη διαφάνεια που είναι ο προπολογισμό 4SP ε, να σας πω ότι εργαζόμαστε σε αυτή την ε, μονάδα από το 2015 ώστε να στηρίξουμε την ε, προπαρασκευή, την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Ήδη το 2015 και 2016 λάβαμε 3 εκατομμύρια για τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Δεν είναι το, σύστημα, το πρόγραμμα μάλλον στήριξης των μεταρρυθμίσεων, αλλά η προπαρασκευαστική δράση για αυτό. Λάβαμε ε, έχουμε να λάβει ε, ε, για την περίοδο 16 μέχρι 20 46,7 εκατομμύρια υπό τον τίτλο 1β. Τίτλος 2 είναι το EFRD. Αυτό Αυτά έχουμε λοιπόν για την ώρα. Έχουμε δεσμεύσει τα κονδύλια για το 2017 και 2018 και τώρα προχωράμε για την υλοποίηση του προγράμματος ε, για το 2018. Να σας δείξω τώρα τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Εδώ έχουμε το ιστορικό για την ε, δαπάνη των κονδυλίων που λάβαμε το 17 και το 2018. Το 2017 καλύψαμε 16 κράτη-μέλη. Είχαμε επιπλέον 271 αιτήσει για 83 εκατομμύρια και δεθήκαμε 159 αιτήματα. Το 2018 είχαμε προπολογισμό 30,5 εκατομμύρια, ενώ είχαμε αιτήματα από, 400, από 24 κράτη-μέλη, 404 αιτήσει για 152 εκατομμύρια και επιλέξαμε 146 αιτήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση στο πρώτο και δεύτερο έτος του προγράμματος. Και ε, όπως γνωρίζετε αυτό προσπαθήσαμε να το τροποποιήσουμε μέσω του ε, τροποποίησης του προγράμματος διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων. Ε, λάβαμε λοιπόν πολλά διαφορετικά αιτήματα υπό ε, στη διάρκεια του 17 και του 18 πολλές αιτήσει. Εδώ βλέπουμε την κατανομή των αιτήσεων ανακράτη-μέλη και την κατανομή των αιτήσεων στις διάφορες, στους διάφορους τομείς πολιτικής. Θα διαπιστώσετε λοιπόν ότι τα περισσότερα αιτήματα προέρχονται, αιτήσει μάλλον προέρχονται από project που θέλουν να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Εδώ έχουμε την κατανομή των επιλεγμένων αιτήσεων για το SRSP. Έχουμε 56% που συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, το 7% συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το 28% συμβάλλει στις προτεραιότητες της Ένωσης και το 9% συμβάλλει προς τα κράτη-μέλη και τις δικές τους προτεραιότητες. Εδώ βλέπετε λοιπόν τι κάνουμε στο πλαίσιο του SRSS και του SRSP τα τελευταία δύο χρόνια. Τώρα θα περάσω στο επόμενο σημείο όπου μου ζητήθηκε να μιλήσω. Κατέβομαι λίγο. SRSP σε σχέση με το ε, μέσο για την ε, επίτευξη των μεταρρυθμίσεων, γιατί υπάρχει ε, αμφισβήτηση για το ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο πρόγραμμα και το εργαλείο επίτευξης των μεταρρυθμίσεων. Καταρχάς έχουμε το πρόγραμμα στήριξης των διαφορετικών αλλαγών. Είναι ένα πρόγραμμα υπό το τρέχον MFF PDP 2014-2020 προσφέρει τεχνική στήριξη στα κράτη-μέλη και πάλι είναι τελείως προαιρετικό. Ε, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα κάτι μέλη να ζητήσουν τεχνική βοήθεια είναι προαιρετικό, επί προαιρετικής βάσης. Αυτό το τμήμα του προγράμματος, δηλαδή τεχνική υποστήριξη, θα συνεχιστεί, υπάρχει πρόταση να συνεχιστεί μετά από το 2020 ως το ε, μέσο για την τεχνική υποστήριξη. Το SRSP όσο έχει σήμερα λοιπόν θα είναι τμήμα ε, του προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Προχωρώ τώρα στην ε, μεταρρύθμιση, ε, μάλλον στο μέσο για την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων. Είναι ένα άλλο μέσο ε, στο πλαίσιο της στήριξης για τις μεταρρυθμίσεις. Είναι το εργαλείο επίτευξης μεταρρυθμίσεων. Έχουμε επίσης την διευκόλυνση για την μετατροπή για να μπορέσουν δηλαδή τα κράτη που δεν είναι ακόμα μέλη της Ένωσης να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να μπουν στην, Ευρω... στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Έχουμε λοιπόν μια πιλωτική φάση που όπως εξηγούμε έχει τη μορφή τροποποίησης στον κανονισμό CPR. Τι είναι λοιπόν αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο που προβλέπει και παρέχει ε, δημοσιονομικά κίνητρα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Και το πιλωτικό πρόγραμμα στόχο έχει να δει πώς θα λειτουργήσει και στο μέλλον. Η ιδέα είναι να δοθούν οικονομικά κίνητρα. Δεν είναι ο στόχος να καλυφθεί το κόστος των μεταρρυθμίσεων, αλλά να δοθεί κίνητρο στα κρατη να προβούν σε, στις μεταρρυθμίσεις αυτές και να τις προωθήσουν. Η πρόταση είναι να συνεχιστεί και μετά από το PDP του 2020. Εάν εγκριθεί η τροποποίηση του CPR, θα μπορούσε να ξεκινήσει η εφαρμογή της πιλωτικής φάσης το 2019, για την περίοδο 2019 με 2020, ώστε να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για το μελλοντικό αυτό εργαλείο, πώς δηλαδή θα γίνει λειτουργικό, πώς θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να υποβάλουν προτάσεις για την μεταρρύθμιση και πώς θα δεσμευτούν Μιλάμε λοιπόν για μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη αναφερθεί από τον ΕΡΙΚ. Πρόκειται και μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στις συστάσεις αναχώρα υπό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, καθώς επίσης μεταρρυθμίσεις που υποδεικνύονται στα συνοδευτικά μέσα και μάλλον έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Δηλαδή, πέρα από τις συστάσεις αναχώρα, περιλαμβάνονται διάφορες προκλήσεις στις εκθέσεις αναχώρα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και μπορεί και αυτό να αποτελέσει τη βάση για την υποβολή προτάσεων μεταρρύθμισης. Καλύπτονται πολλές, πολλοί τομείς λοιπόν και Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα εξ αυτών που τα κάνουν τα κατημέλη είναι το να κάνουν ένα πρόγραμμα εγγύησης με εισοδημάτων. Ε, εμείς λοιπόν το σχεδιάζουμε και, και γίνεται μια πρόταση για την εφαρμογή του. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει καταρχάς τον σχεδιασμό του προγράμματος ε, ένα πιλωτικό, ένα σχέδιο, δοκιμαστικό δηλαδή, και μετά εφαρμογή του. Αυτό είναι ένα παράδειγμα λοιπόν μπορώ να σας δώσω, αλλά μπορώ να σας δώσω και ένα σωρό άλλα διαφορετικά παραδείγματα για πιθανές ε, ε, μεταρρυθμίσεις που μπορεί να αφορούν πολλούς τομείς. Αυτό εδώ αφορά το κοινωνικό τομέα. Θα μπορούσαμε να έχουμε παραδείγματα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σε κάποια κράτη-μέλη υποστηρίζονται η λειτουργική αναδιοργάνωση των νοσοκομείων, για παράδειγμα. Ε, αυτό είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη προωθούν ε, αλλαγές στην αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, των δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να είναι μεγάλου φάσματος μεταρρύθμιση σε πολλά κράτη-μέλη. Υπάρχουν δηλαδή ένα σωρό μεταρρυθμίσεις που μπορεί να καλυφθούν εδώ ή μπορεί να προταθούν. Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο και είναι κάτι που έχουμε μάθει από την λειτουργία των διαστατικών προγραμμάτων είναι πολύ σημαντικός ο διάλογος, ο διάλογος που γίνεται εκ των προτέρων ανάμεσα στα κρατημέλη και την Κομισιόν, έτσι ώστε στο πλαίσιο της τεχνικής μας υποστήριξης έχουμε εντατικούς διαλόγους πριν να υποβληθεί η πρόταση ε, για στήριξη. Το ίδιο γίνεται και στο πλαίσιο της υποβολής δεσμεύσεων περί μεταρρυθμίσεων, όπου τα κράτη-μέλη εμπλέκονται σε θετικό διάλογο για τη φύση της δέσμευσης που αναλαμβάνουν για μεταρρυθμίσεις και έτσι ε, μπορεί να έχουν εξομαλυνθεί πολλά προβλήματα εκ των προτέρων, πριν να υποβληθεί καν η πρόταση και να έχουν έτσι διευκρινιστεί και οι λεπτομέρειες πριν να υποβληθεί καν επισήμως η πρόταση. Δεν θα καταναλώσω άλλο το, χρόνο σας, θα σταματήσω σε αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ενδεχόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό μου θύμισε και τη συζήτηση που είχαμε για την πρώτη πρόταση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αν θυμάστε καλά, αυτή η Επιτροπή ήταν το μέρος όπου ξεκίνησε η όλη η συζήτηση. Και τώρα μιλάμε για το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και το αποθεματικό επιδόσεων. Ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, θεωρούμε πως ε, είναι κάτι που χρειαζόμαστε και στηρίζουμε ε, το όλο εγχείρημα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο μεγάλη μου χαρά στον κύριο Σπύρο Σπυρίδων, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΚΟΤΕΡ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών για την ε, αλλαγή ε, του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ε, κύριε Σπυρίδων, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να μιλήσω εκ μέρου τη Επιτροπή των Περιφερειών για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και την τροποποίηση αυτού. Θα ήθελα ε, να μιλήσουμε λοιπόν για τη στήριξη των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να μεταφέρω τις θερμέ ευχές του Προέδρου της Επιτροπής Κοτέρ, κ. Όσφαλτ, και των πρόσφατα διοριστέντων ε, εισηγητών, κ. κατιουσκα Μαρίνη και ε, Μίχαλ Σνάιντα. Μετά τη γνωστοποίηση της πρότασης της Κομισιόν το Δεκέμβριο πέρυσι, η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να εγκρίνει ένα ψήφισμα την πρώτη ολομέλειά της το 2018. Επομένως, την 1η Φεβρουαρίου του 2018, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ολομέλειά της ενέκρινε ψήφισμα το οποίο καθαρίζει τη θέση της όσον αφορά τη χρήση του αποθεματικού επίδοσης για τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις και δείχνει την θέση της Επιτροπής των Περιφερειών σε ό,τι αφορά τη χρήση του αποθεματικού για τις ε, μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τώρα τα κύρια σημεία του ψηφίσματος ε, εν συντομία. Καταρχάς, ε, κάποια σημεία από προηγούμενες γνωμοδοτήσεις Επιτροπής των Περιφερειών. Έχουμε τονίσει εδώ και καιρό ότι δεν πρέπει να τιμωρούνται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές κάποιων κρατών μελών ε, διότι υπήρξαν προβλήματα λοιπού εφαρμογής οικονομικών πολιτικών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσιονομικών ελλημάτων. Επίσης, ήμασταν αντίθεση, αντίθετοι ε, στην υποταγή της ε, πολιτικής ε, συνοχής, μια που η πολιτική αυτή είναι από, αυτόνομη και προκύπτει από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Επίσης, σε ό,τι αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020, τονίζουμε ότι το μέλλον της πολιτικής συνοχής στα προγράμματα εθνικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να διατηρεί την τοπική διάσταση και την αποκεντρωμένη προσέγγιση της ε, εταιρικής σχέσης. Επίσης, με βάση αυτούς τους συλλογισμούς είμαστε υπέρ της προώθησης οικονομικής και κοινωνικής συνοχής ως έναν στόχο για όλες τις πολιτικές. Μια από αυτό απορρέπονται συνθήκες. Ε, η πολιτική συνοχή, λοιπόν, όπως προκύπτει από τις συνθήκες, δεν καθίστε υποχρέωση ε, ε, στα κράτη-μέλη να διεξάγουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, απορρίπτουμε την επιχειρηματολογία συμμόρφωσης ε, με τις αρχές του κανονισμού περικοινών διατάξεων, διότι ο στόχος της πολιτικής συνοχής δεν είναι να στηρίξει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη, αλλά να μειώσει τις ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών εις βάρος των ε, λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής, σε παραβίαση των αρχών της συγχρηματοδότησης και της επιμερισμένης διαχείρισης. Οι αρχές αυτές είναι ζωτική σημασία για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τη ε, ανάληψη ευθυνών ε, σε ό,τι αφορά τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και τη χρηστή διακυβέρνηση, καθώ και τη μεγιστοποίηση ε, τη μόχλευση τη πολιτική συνοχή. Επίση, τονίζουμε ότι στο πλαίσιο της ε, αρχής της πολυεπίπεδης ε, διακυβέρνησης, η χρήση των ε, Ευρωπαϊκών Διευθυντών και Επενδυτικών Ταμείων για σκοπό τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων απαιτεί δράση συντονισμένη σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς αυτό δεν επιτρέπεται στην πρόταση της Επιτροπής. Επιπλέον, διαπιστώνουμε μία αντίφαση μεταξύ της χρήσης των ε, πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για τη χρηματοδότηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη και με την υποχρέωση της θεματικής συγκέντρωσης όπως ορίζεται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Επίσης, ανησυχούμε για την ε, χρονική στιγμή της πρότασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα εργαλείο για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και επίσης πρότεινε να χρησιμοποιήσουμε το αποθεματικό επιδόσεων για τη χρηματοδότηση ενός ε, νέου ε, μέσου υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων χωρίς να έχουν ε, παρουσιαστεί οι λεπτομέρειες της πρότασης. Τώρα που έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα επιμέρους στοιχεία του, μπορούμε να δούμε βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες και να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτό όμως δεν μας έχει κάνει να αλλάξουμε άποψη για την παρούσα πρόταση της Επιτροπής. Επίσης, σημειώνουμε ότι η, ο λόγος ύπαρξης του αποθεματικού επιδόσεων είναι να στηρίξει τις προτεραιότητες εκείνες που πραγματικά το αξίζουν. Ωστόσο, η πρόταση χρήσης τους θα αποθαρρύνει τις ε, περιφέρειες και τις αρχές ε, διαχείρισης. Επίσης, ε, ανησυχούμε για, το, για τη χρονική στιγμή της πρότασης αυτής που μπορεί να οδηγήσει σε νομική ανασφάλεια και καθυστερήσεις είναι πολύ ε, κρίσιμη η χρονική στιγμή την οποία διανύουμε. Και η πρόταση ε, της Επιτροπής δεν μπορεί να ε, συνδυαστεί χρονικά με τις άλλες προτάσεις που έχουμε ήδη υποβληθεί. Με, για την περίοδο μετά το 2020, η παρούσα πρόταση λοιπόν δεν βασίζεται σε πρώτερη εμπειρία μας. Η πρόταση να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ταμεία για τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων βασίζεται στους στόχους της πολιτικής συνοχής και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη έχει ε, αναφερθεί από το πρόγραμμα στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τα προγράμματα τεχνικής ε, υποστήριξης του ε, Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να... Ε, λάβουν πρόσθετη στήριξη από εθνικά προγράμματα και από διάφορα προγράμματα τεχνικής υποστήριξης. Επομένως, η Επιτροπή των Περιφερειών με την έγκριση του ψηφίσματος αυτού στην Ολομέλεια της 1ης Φεβρουαρίου αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή των Περιφερειών Δηλώνει μάλιστα να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που έχει να αμφισβητήσει την νομοθετική πράξη αυτή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλου αριθμός 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σε ό,τι αφορά τι προτάσει για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε λεπτομερή συζήτηση για την πολιτική συνοχή, για τι Ευρωπαϊκέ μεταρρυθμίσεις και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θεωρούμε ότι η πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την οικονομική ε, και κοινωνική βιώσιμη διακυβέρνηση αποτελεί προαπαιτούμενο. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Σπυρίδων. Αυτή ήταν η θέση της Επιτροπής των Περιφερειών. Because of the special request of the members of Κατόπιν ειδικού αιτήματο των μελών της ΡΕΤΖΙ, έχουμε και εκπροσώπους του ελεγκτικού συνεδρίου, τους οποίους καλωσορίζω. Ο κύριος Γκέρχαρντ Ρος, διευθυντής ε, του τμήματος 1 και κύριος Πρόκοπ, Ελπίζω να προφέρω σωστά τα ονόματά σας. Από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Παρακαλώ. Ε, thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε τις παρατηρήσεις ε, και τα συμπεράσματά μας ε, για το αποθεματικό επίδοσης στο πλαίσιο της περίοδου 14-20 βάσει της πρότασης της μεταβίβασης τελείων από το ένα στο άλλο. Δεν υπάρχει ακόμα γνωμοδότηση του Ελληνικού Συνεδρίου. Θα κάνω λοιπόν μερικά γενικά σχόλια με βάση την ε, εμπειρία του παρελθόντος. Το Ελληνικό Συνέδριο έχει καλύψει το αποθεματικό ε, επιδόσεων ε, και στο παρελθόν σε μια σειρά περιπτώσεων. Όταν προτάθηκε το νομικό πλαίσιο, εμείς κάναμε μια γνωμοδότηση. και σε δύο κεφάλαια στην ετήσια έκθεση του 2013 και του 2014. Και υπήρχε ήδη στο υιοθετημένο ε, πλαίσιο επιδόσεων. Μετά είχαμε και με ειδική έκθεση για την εξάντερη αιρεσιμότητα και το παθηματικό επιδόσεων του 2017. Αυτές είναι οι εκθέσεις μας. Λοιπόν, ας διατρέξω τα βασικά συμπεράσματά μας και παρατηρήσεις μας. Στην γνωμοδότηση ε, του 2011 λέμε ότι το πλαίσιο συνοχής βασίζεται πολύ ε, στους πόρους που εισάγονται, στο input και όχι αρκετά στις επιδόσεις. Ένα, μια καλή κίνηση προόδου θα ήταν το αποθεματικό ε, επιδόσεων. Και γι' αυτό Είπαμε όμως ότι ο σχεδιασμός ενέχει τον κίνδυνο να επικεντρώνεται πιο πολύ ε, στα κονδύλια που δαπανώνται και όχι τόσο στα αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα από τα ζητήματα που είχαμε θίξει. Άλλο, για να λειτουργήσει σωστά το παθηματικό, λέγαμε ότι θα πρέπει ε, να γίνει σωστή στάθμιση των στόχων, να είναι δηλαδή αρκετά φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική παράλληλα. και ότι αυτό θα είναι το κλειδί της επιτυχίας, είχαμε πει τότε. Και τέλος, η κατανομή του αποθεματικού επιδόσεων θα πρέπει ε, να υπόκειται και σε επαρκή επίπεδα υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Θα έχουμε έκθεση για την απορρόφηση τον Οκτώβριο, όπου θα σταθούμε ακριβώς στην περίοδο και για το 7-13 και για το 14-20. Μετά, μερικά χρόνια αργότερα, είπαμε ότι με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται το αποθεματικό, μάλλον δεν θα έχει ε, σημαντικά αποτελέσματα, θα έχει μόνο οριακά ε, αποτελέσματα. η συμπερίληψη των οικονομικών δικτών ενέχει τον κίνδυνο της αντιστροφής του σημείου εστίασης προς την απορρόφηση και όχι προς τις επιδόσεις. Και είπαμε ότι για να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά το αποθεματικό, αυτό θα εξαρτηθεί κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τους ε, στόχους, ε, κατά πόσο έχουν επιτευθεί εγκαίρως ε, και με τον σωστό τρόπο. Είχαμε λοιπόν επισημάνει κάποιους κινδύνους. Το 2017 εκδώσαμε μια ειδική έκθεση για την εξάντερεσιμότητα και το αποθεματικό επιδόσεων. Για το αποθεματικό είπαμε το ποσό ήταν 20 δις ευρώ, σημαντικό ποσό για ένα αποθεματικό και καταλήξαμε στο συμπέρασμα, όπως και στο παρελθόν, ότι ήταν πολύ μικρό το κίνητρο ε, για καλύτερα αποτελέσματα, δεν υπήρχε σωστός γιατί τα βασικά στοιχεία ήταν το input και το output. Τι βάζουμε και τι αποτελέσματα έχουμε. Ε, και ότι μάλλον δεν θα υπήρχε σημαντική ανακατανομή των κονδυλίων και των δαπανών προς ε, καλύτερα προγράμματα. Βέβαια υπάρχουν και δυνατά σημεία ε, του υποθεματικού. Βρήκαμε δείκτες που προκύπτουν από την λογική της παρέμβασης. Έτσι, εξορισμού θα πρέπει να συνδέονται με τους στόχους. Οι στόχοι ε, τίθενται εκ των προτέρων και κατόπιν συμφωνίας με τα κράτη-μέλη. Αντίστοιχα εγχειρήματα είχαμε κάνει και το 2000 με 2006 και στην πραγματική περίοδο 2007-2013. Μία από τις βασικές αδυναμίες όμως ήταν αυτή η έλλειψη ανατολισμού. Είχαμε αναλύσει δείκτες που είχαν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο επιδόσεων και είδαμε ότι το 57% αφορούν μόνο τα αποτελέσματα output. Μόνο το 1 τρίτο αφορά το input, ε, τι δαπανούμε και μόλις 0,3% αφορούσε πραγματικά τα αποτελέσματα. εφόσον παραμένει εντός του προγράμματος, το αποθεματικό και εντός του φακέλου των κρατών μελών, υπάρχει ε, πάντα ανταγωνισμός για τα ε, προγράμματα με, τα καλύ... με τις καλύτερες επιδόσεις. είπα ότι θα πρέπει να τίθενται σωστοί στόχοι και φιλόδοξοι και ρεαλιστικοί παράλληλα. Αναλύσαμε τους δείκτες και βρήκαμε ότι το 46% των δεκτών ήταν δύσκολο να διαπιστώσουμε κατά πόσο ήταν ρεαλιστική και φυκτοί. Και η υπαρκτή δυνατότητα αναστολής για τους ε, στόχους που δεν επιτυγχάνονται ε, είναι μάλλον απίθανο να εφαρμοστούν και να επιβληθούν. Είχαμε πει λοιπόν ότι η νομοθετική πρόταση για μετά το 2020 ε, θα πρέπει να, ε, έχει, να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και έτσι να κατανέμονται τα κονδύλια. Τώρα ξέρουμε ότι έχει καταργηθεί το αποθεματικό επιδόσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο και Αυτό θεωρούμε ότι είναι κρίμα γιατί θα μπορούσε να αυξήσει την εστίαση στις επιδόσεις αυτό το μέσο. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για, τις, για τη στήριξη διευθυντικών μεταρρυθμίσεων, εμείς εκδώσαμε γνωμοδότηση το 2017 για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και εκεί είχαμε πει ότι είμαστε υπέρ ε, των πληρωμών βάσει της πλήρωσης ε, προϋποθέσεων ή ε, βάσει της επίτευξης αποτελεσμάτων. Βέβαια, η επιτυχία ενός τέτοιου καθεστώτος εξαρτάται από τη σωστή εφαρμογή. Κάποια ερωτήματα που θέτουμε τώρα εμείς. Τα κονδύλια που μετατίθενται από το παθηματικό επιδόσεων συμβάλλουν ακόμα στους στόχους της πολιτικής συνοχής. Υπάρχει δυνατότητα να ταυτοποιήσουμε τέτοιους ε, στόχους και βασικά στοιχεία που μας ε, βοηθούν να μετρήσουμε την πρόοδο και αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων. Πώς αξιολογούμε λοιπόν ε, και πώς θεωρούμε ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Ποιος παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία, ποιος την ελέγχει όταν γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Μετά, αυτή η διάρκεια των τριών ετών σαφώς και περιορίζει ε, το είδος των μεταρρυθμίσεων που μπορούν ε, να προχωρήσουν. Μένω εδώ και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτές τις παρουσιάσεις είχαμε σήμερα με τις επιμέρους θέσεις. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση ξεκινώντα από τους ε, συνεισηγητέ, που είναι και συντονιστές, η κυρία Κρέλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μισό κομμάτι της ακρόασης ε, αναφέρεται σε θέματα τα οποία δεν θέλαμε καν να θίξουμε σήμερα διότι σήμερα το μόνο που θέλαμε να συζητήσουμε είναι αν η πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι κάτι το οποίο ε, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε. Δεν τίθεται θέμα ε, του αν θεωρούμε καλό ή όχι το μέσο, δεν τίθεται θέμα του αν θεωρούμε καλό ή όχι το αποθεματικό επιδόσεων. Αυτά είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό που μας μένει, αν τα αφαιρέσουμε αυτά, είναι η πρόταση του κυρίου Φανμπρέσκα, η πρόταση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η θέση του Συμβουλίου, το οποίο είναι αντίθετο, και η θέση της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία επίσης είναι αντίθετη στην πρόταση της Επιτροπής. Και ως εισηγήτρια, ως συνεισηγήτρια μάλλον, κατέστησε σαφέ από την αρχή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποτέ δεν ήθελε ένα αποθεματικό επιδόσεων, διότι δεν θεωρεί πως ε, κάτι τέτοιο είναι ε, σωστό στην προκειμένη περίπτωση, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς. Είμαι κάθετα αντίθετη στο να ε, παίρνουν χρήματα από την πολιτική συνοχή για να στηρίξουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όποιες και αν είναι αυτές. Και στο μεταξύ Συζήτησα αρκετά με διάφορους ενδιαφερομένους φορείς ε, και άκουσα ότι υπάρχουν χώρες, ε, η Πορτογαλία συγκεκριμένα, που ε, ενδιαφέρεται για την υλοποίηση τέτοιων πιλωτικών προγραμμάτων και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες διαβουλεύσεις χρειάζονται ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις επιμέρους περιφέρειες, ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να ξεκινήσει απλά ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και αυτό μόνο για την περίοδο 2019-2020. Μόνο για τον ένα χρόνο λοιπόν, γιατί μετά έτσι κι αλλιώς τελειώνει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το ε, έχω ξαναπεί. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πρέπει να γυρίσει πίσω από εκεί που ήρθε για να προλάβουμε οποιασδήποτε ζημιές. Και γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει ορισμένα, ορισμένες περιπτώσεις που μπορούν να θεωρηθούν προηγούμενο. Ήδη υπάρχουν ορισμένα πιλωτικά προγράμματα τα οποία έχουν ε, υλοποιηθεί. Αλλά εάν ε, πραγματικά έχετε κάτι τέτοιο, σας παρακαλώ να το εφαρμόσετε. Δεν χρειάζεται να αλλάξει ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων. Μπορείτε να κάνετε κάτι δοκιμαστικό στην αρχή πρωτού πάτε σε τόσο δραστικές αλλαγές ε, που θα κοστίσουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Διότι ξέρετε ότι όταν ξεκινήσει κάτι από ένα για μέλος μετά θα υπάρξουν αντιδράσεις από πολλά και στο τέλος δεν θα μείνει δεκάρα για την πολιτική συνοχή αν ο καθένας παίρνει κατά το δοκούν. Μετά το 2020, αν θέλουμε να συζητήσουμε το μέλλον της πολιτικής συνοχής, ε, τότε ε, μπορούμε να το δούμε αλλιώς ε, με τον συνεισηγητή κύριο Νόβακοφ ε, συμφωνούμε απόλυτα για το ότι πρέπει να δούμε το ενδεχόμενο του, ε, της κοινή διαχείρισης και της κοινή ανάληψης ευθύνης στην στήριξη των διαθερωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτό να το κοιτάξουμε. Αλλά δεν θεωρώ πως αυτή τη στιγμή έχουμε την δυνατότητα να προβαίνουμε σε τόσο δραστικές αλλαγές. Γι' αυτό λοιπόν άσκη κοιτάξουμε ε, λίγο προς τα πίσω και ας δούμε τι έχει γίνει ε, στα λίγα πιλωτικά προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται να ε, πάρουμε 20 δισεκατομμύρια ευρώ και να αλλάξουμε τα πάντα. Ας διοργανωθεί λοιπόν ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην Πορτογαλία, όμως χωρίς αποθεματικά επιδόσεων και όλα αυτά που προτείνεται. Νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα έπρεπε πραγματικά να αποσύρει την πρότασή της, διότι γνωρίζετε ότι υπάρχει και η πρόταση περί καλύτερης νομοθεσίας και θα ήθελα να σας παραπέμψω σε αυτή. Okay. It was the position of Ωραία. Αυτή ήταν η θέση της μίας συνεισηγήτριας. Ο κύριος Βανίστελ Ρόιν. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να σας δώσω μια άλλη λύση. Ε, από την αρχή, ως συνεισηγητές, ήμασταν ιδιαίτερα δραστήριοι. Και ο Επίτροπος είχε έρθει εδώ και είχαμε πλήρη συζήτηση για το νέο μέσο και τη μορφή που θα πάρει μετά το 2020 τι θέση θα έχει. Θα έχει ξεχωριστό προπολογισμό, θα συνδέεται με την ε, πολιτική συνοχή. Εν τω μεταξύ έχουμε την απάντηση, έχουμε ένα νέο ε, προπολογισμό για τις τριθωτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν θα αφαιρείται πια από τα διαρθρωτικά ταμεία. Είχαμε λοιπόν μια συνολική συζήτηση για αυτό το αποθεματικό επιδόσεων και μήπως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλα αποτελέσματα, ποια είναι η πρόθεση της Επιτροπής. Είχαμε προφορικό ερώτημα στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Με πολύ σαφή ερωτήματα από την Επιτροπή Ρέτζι. Βάσει και των όσων είπαμε στην έκθεση της κυρίας Βέστφαλ για τα building blocks, ότι αν τα κράτη-μέλη κάνουμε περισσότερες δαπάνες, τότε το αποθεματικό επιδόσεων μπορούν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νωρίτερα. Και θέλαμε να δούμε ποια είναι και η γνώμη και η απάντηση της Επιτροπής. Γι' αυτό θέσαμε αυτά τα ερωτήματα και πήραμε σαφέστατες απαντήσεις. Να τη διαβάσω την απάντηση. Η Επιτροπή δεν είναι διατεθειμένη να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή ε, στην τρέχουσα νομοθεσία, στην ισχύουσα νομοθεσία. Και εδώ έχουμε μία αλλαγή. Παραθέτω, έτσι. Γιατί, πρώτον, θεωρούν ότι σε ένα κράτος μέλος όλοι οι δείκτες στο πλαίσιο επιδόσεων θα πρέπει να αποφασίζονται με βάση και τις ισχύουσε νομικέ διατάξεις. Αυτό είναι το πρώτο και ισχύει. Το δεύτερο που λένε. Και αυτό ισχύει μέχρι το τέλος του 2019. Λένε ότι αυτό περιπλέκει το σύστημα, θα περιέπλεκε το σύστημα και θα αύξανε το άχθος για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες χωρίς αυτά αποτελέσματα και ωφέλη. Ορίστε, ξεκάθαρη η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λένε ότι θέλουν να ακολουθήσουν την ισχύουσα νομική βάση. Και τώρα η ίδια Επιτροπή, γιατί ενιαία είναι η Επιτροπή στις επιδόσεις της, ξαφνικά παίρνουμε μια κατά τη διαφορετική πρόταση. Και θυμάμαι ότι στην αγόρευσή μου είχα πει ότι χρειάζεται ευελιξία και από τις δύο πλευρές αν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Ήθελα να δω τι περιθώριο ευελιξίας υπάρχει. Και είπα ότι αν δεν δώσετε περισσότερη ευελιξία, δεν θα υπάρξει πρόοδος. Αυτό είναι το συμπέρασμα που έχουμε τώρα και αυτό που είπε η κυρία Κρέλ. Και το είπε η κυρία Μακάρθη ξεκάρθα. Δεν ήταν αυτή η αφετηρία. Ξεκινήσαμε από μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία και εμείς ως συνεισηγητές είπαμε ναι ε, στο πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων. Και τώρα η κυρία Τόμασιτς νομίζω θα, σύντομα θα παρουσιάσει την πρότασή της στην Ολομέλεια. για την επόμενη αυτή διαδικασία στήριξης. Επομένως, υπάρχει δυνατότητα. Ο κύριος Βανμπρέσκα σήμερα ξεκίνησε νωρίς, από τις 9 το πρωί, όπως και εμείς. Και μας μετέφερε το μήνυμα. το αποθεματικό επιδόσεων, το οποίο βέβαια τελικά δεν θα υπάρχει στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Κάπως ε, θα αποδημήσεις κύριον ε, και νωρίς αυτό το μέσο. Δεν ε, υπάρχει όρεξη και βούληση από το Συμβούλιο. και η Επιτροπή των Περιφερειών να παρουσίασε τα επιχειρήματά της. Ίσως μπορούμε να λάβουμε και από το ελεκτικό συνέδριο όλα τι διαφάνειες, γιατί εγώ δύο βρήκα μόνο και το ζουμί ήταν ε, μεταξύ αυτών των δύο. Το μοναδικό συμπέρασμα είναι αυτό το ερώτημα που κάνατε. Είτε να αποσυρθεί η πρόταση, είτε να ψηφίσουμε τον Ιούλιο όπως κάναμε στην ε, ΙΜΚΟ. Απλώ να καταψηφίσουμε και πάει η πρόταση από πλευρά Κοινοβουλίου. Και μετά η Επιτροπή μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να μιλάει. Ποιο ξέρει. Μπορεί να ακολουθήσει τη δική σας ε, πρόταση. Ορισμένες χώρες να βγουν μπροστά. η διασύνδεση εδώ με το αποθεματικό επιδόσεων δεν είναι αυτή που θέλαμε εμείς. Δεν ήταν απλώς ένα βήμα παραπέρα. Εντάξει, τα πρώτα βήματα μας βρήκαν σύμφωνους. Και οι ειδικέ αναχώρα συστάσει συνδέονται με την ε, υλοποίηση των προγραμμάτων. Εντάξει, οπότε δεν είναι και κάτι το απολύτως εξωφρενικό. Προτείνω λοιπόν είτε να αποσύρει η Επιτροπή σήμερα ή αύριο την ε, πρότασή της, είτε να προετοιμάσουμε ε, την ε, ψηφοφορία στον Ιούλιο. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πράγματα. για τις παρουσιάσεις θα διανεμηθούν στα μέλη της Επιτροπής μας όλες ε, οι παρεμβάσεις και παρουσιάσεις. Όσο ήθιστε μετά το τέλος της συνεδρίασής μας και της πρωινής συνεδρίασης και της απογευματινής. Θα τα λάβετε λοιπόν. Δεύτερον, το πρωί κάτι λέγατε για τις πίτες που ανέφερε ο πρόεδρος, ε, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Τώρα εμένα δεν μου αρέσει αυτή η νήξη που κάνατε για τις ε, κηδείες και την αποδίμηση κύριων. Α, ζητώ συγγνώμη. Ούτε κομμάτι της πίτας πήρα όμως. Ούτε εγώ την κηδεία, λέει η Πρόεδρος. Κυρία Τόμασιτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. καθότι παρόλο που ε, δεν είμαστε υπέρ της, ε, των μεταρρυθμίσεων αυτών, θα ήθελα επί τη ευκαιρία να εκφράσω την στήριξή μου προς αυτή την πρόταση, γιατί χρησιμοποιείται ως πραγματικό κίνητρο για ορισμένα κράτη-μέλη που χρειάζονται τέτοιες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, στην υγειονομική περίθαλψη, νοσοκομεία, στο δημόσιο τομέα ένα παράδειγμα των βασικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Δυστυχώς μέχρι τώρα κάποια κράτη-μέλη δεν είχαν ε, ε, την τεχνογνωσία ή την απαραίτητη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, προβούν σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει διάλογος μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής και αυτή η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να είναι μια καλή αφετηρία και φυσικά ξέχασα να πω ότι πρέπει να ευθυγραμμίσετε με την πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ κύριο Βαν Μίλτενμπουργκ. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτή η πιο θετική προσέγγιση ε, από πλευρά ECR ε και εμεί συμφωνούμε ότι υπάρχει σαφή σύνδεση, ε, ανάγκη ε, διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και πολιτική συνοχή. Εδώ έχουμε το καλύτερο δυνατό επενδυτικό κλίμα. Αυτό για μα είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια μετά τίθενται μια σειρά ερωτημάτων ε, για την υλοποίηση. Και νομίζω ότι το νόημα της σημερινή ακρόασης αυτό είναι, να θέσουμε ερωτήματα. Γιατί δεν το έπραξαν οι συνεισηγητές. Εγώ έχω ερωτήματα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς το Ελληνικό Συνέδριο, για παράδειγμα. Ένα ερώτημα που ήδη έφυξε προηγουμένως είναι πώς ε, ορίζουμε τα ποσά που θα πρέπει να θεωρηθούν ως ποσό που αποτελεί κίνητρο, δεν συνδέεται με, με το κόστος. Αλλά πώς γίνεται αυτό, με ποια κριτήρια, είναι ένα καταποκοπήν ποσό, πώς προσδιορίζεται. Μετά, κάτι που ακούστηκε στο τέλος ε, από το ελεγκτικό συνέδριο. Εγώ είμαι υπέρ τη αξιολόγηση και της επιτυχούς ε, υλοποίηση των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Αλλά πώς μπορούμε να την αξιολογήσουμε, Πότε λέμε ότι ήταν επιτυχή η υλοποίηση. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε κριτήρια. Και εκεί τίθεται το θέμα της λογοδοσίας. Ακόμα λοιπόν δεν είμαι σίγουρος πως όλα αυτά θα γίνουν στην πράξη. Είμαι λοιπόν θετικά διακείμενος ως προς το ευρύτερο σκεπτικό και θεωρώ ότι είναι καλό να αρχίσουμε τους πειραματισμούς αλλά πρέπει βέβαια να απαντήσουμε και τέτοια ερωτήματα. Δεν γίνεται το Κοινοβούλιο να συμφωνήσει επί μίας πρότασης όταν σε μερικά χρόνια μπορεί να έχουμε πρόβλημα με το ελεγκτικό συνέδριο και να μας λέει συμφωνήσατε και εγκρίνατε έναν μηχανισμό όταν ακόμα παραμένουν ε, ανοιχτά ζητήματα, Ιδίω ε, στη λογοδοσία. Είμαστε αιρετοί εκπρόσωποι, λογοδοτούμε στους ε, ψηφοφόρους μας ιδίως ό,τι αφορά την ε, σωστή χρήση των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων, που είναι χρήματα των φορολογουμένων. Δεν είμαι λοιπόν αρνητικός, απλώς ακόμα με προβληματίζει η πρακτική εφαρμογή όλων αυτών. Ιδίω για τον προσδιορισμό των ποσών, τη πρακτική εφαρμογή, των κριτηρίων και ούτω καθεξή. Χρειάζομαι περισσότερε πληροφορίε πριν μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ε, στο ιστορικό της ομάδας των φιλελευθέρων και καταλήξουμε σε μια επίσημη θέση. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα έχει έρθει η ώρα για συζήτηση και για τις ερωτήσεις φυσικά. Διακόπτω κύριο Νίστελ. Ε, έχετε διαπιστώσει για το αν πράγματι η νομική βάση, σύμφωνα με αυτό που μας είπε και ο Επιτροπός Δομπρόσκης, είναι διαφορετική ε, και ποιο, ποια επιτροπή θα αρμόδια. Τώρα νομίζω η αρμόδια επιτροπή είναι η ΕΚΟΝ. Μας πήρε την ε, αρμοδιότητα, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν αλλάξει οι ρόλοι. Προτού μπούμε δηλαδή σε λεπτομέρειες και μετά καταλήξουμε να γνωμοδοτούμε απλά για έκθεση της Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ. Νομίζω πως έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουμε και όπως είπατε και εσείς συμπερασματικά, τώρα μας μένει το τελευταίο βήμα, το οποίο δεν μπορεί να γίνει ακόμα για τους λόγους που ακούσαμε όλοι. Ναι, φυσικά, ο τελικό χρήστη όμω, ο οποίο μπορεί να είναι ένα κράτο μέλο, αυτό δηλαδή που θα χρησιμοποιήσει τι ε, διαρθρωτικέ ε, μεταρρυθμίσει, ε, θα βρεθεί ενώπιον ζητήματο αρμοδιότητα. Και αυτά είναι εσωτερικά θέματα το ζητούμενο εδώ είναι η στήριξη και αυτό, σε αυτό αποσκοπεί η πρόταση, δηλαδή να στηρίξει τα κρατημέλη που θέλουν να προβούν σε διαρθωτικέ μεταρρυθμίσει. Το ερώτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αν θα δεχτεί ή όχι ε, την ενεργοποίηση μέρου του αποθεματικού επιδόσεων και για ποιου σκοπού, οι οποίοι θα βασίζονται σε ποια κριτήρια. Ε, θα δώσουμε λευκή επιταγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι θέλει ή θα αναλάβουμε το ρόλο ε, του επόπτη για να δούμε πού πηγαίνουν τα χρήματα των φορολογούμενων. Ε, δεν είναι το θέμα, πιστεύω, εδώ ποια επιτροπή θα είναι η καθήλυνα αρμόδια. Μπορεί και να είναι η ΕΚΟΝ. Νομίζω η ΕΚΟΝ θα είναι. Νομίζω πω σε τελική ανάλυση έχουμε υποχρέωση απέναντι στα κράτη-μέλη ε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μισάλη. Μίχελς. Μίχελς. Μάλιστα, νομίζω ε, και εγώ έχω την ίδια άποψη για διαφορετικούς όμως ε, λόγους. Όπως είπε και η κυρία Κρέλ, συμφωνώ μαζί της, ε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε ανάγκη μεταρρυθμίσεων όταν δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Μέχρι στιγμής μόνο ένα κράτος μέλος υπάρχει το οποίο χρειάζεται αυτή την στήριξη όπως ακούσαμε. Ε, γι' αυτό δεν νομίζω πως ε, πρέπει να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις ε, για μόνο μία μεμονωμένη περίπτωση. Έπειτα, ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Το Συμβούλιο είναι κατά. Η Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία βασικά είναι και η αρμόδια και ο αποδέκτης της πολιτικής μας αυτής, είναι αντίθετη για τους ε, ίδιους λόγους και ακόμα περισσότερους και ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει και εδώ κάποια ε, άποψη που συμφωνεί με την Επιτροπή. Επίσης δεν νομίζω πως έχουμε εξετάσει όλες τις παραμέτρους και δεν είναι και τόσο εύκολο να πετάξουμε τις 22 δισεκατομμύρια. Δεν είναι φραγκοδίφραγκα αυτά για να τα δώσουμε έτσι ε, αβίαστα και το θεωρώ ανεύθυνο να σας πω την αλήθεια ε, και με εξοργίζει αυτή η ανευθυνότητα από μέρους Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βάνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη και εγώ συμφωνώ απόλυτα με ε, την προλαλή σας αλλά και με την κυρία Κρέλ. Διαφωνούμε κάθετα με την πρόταση της Επιτροπής για το αποθεματικό επιδόσεων και με την πρόταση να μεταφερθούν πάλι κονδύλια από, τα, από την πολιτική συνοχή σε ένα νέο μέσο. Και δεν διαφωνούμε επειδή θεωρούμε το αποθεματικό επιδόσεων ε, ε, κακό, ούτε επειδή είμαστε αντίθεση, αντίθετοι με την στήριξη των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων ως τέτοια. Ο λόγος που δεν θέλουμε τη συγκεκριμένη πρόταση είναι, όπως υπόθηκε και από τους ε, προηγούμενους συναδέλφους, επειδή δεν τη χρειαζόμαστε. Υπάρχει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο παρουσιάστηκε στις 2 Μαΐου. Υπάρχει νέα γραμμή του προϋπολογισμού ε, για διάφορα μέσα της ε, Νομισματικής Ένωσης και αυτά, ε, αυτό εδώ είναι ένα νέο μέσο με θικιά του γραμμή προϋπολογισμού. Πολλά τα λεφτά, όπως είπατε και εσείς, και δεν είναι δίκαιο για τις περιφέρειες, είναι ε, απογοήτευση να περιμένουν κάτι και να μην ε, ε, έχουν αποτέλεσμα, να μην τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Και θεωρώ λοιπόν ε, και εγώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποσύρει την πρότασή της. Η κυρία Νταμάτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, είμαστε ενώπιον μιας τροποποίησης του κανονισμού για τις κοινέ διατάξεις και έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο να θελήσει να δώσει μια κατεύθυνση τέτοια η Κομισιόν στην πολιτική συνοχή, αφαιρώντας όμως και άλλα κονδύλια. Ακούσαμε από το Συμβούλιο ότι είναι κατά και την Επιτροπή των Περιφερειών ότι είναι κατά και από ό,τι κατάλαβα και το μεγαλύτερο τμήμα αυτής μας της Επιτροπής είναι επίσης κατά. Αυτή την πρόταση λοιπόν που συζητάμε σήμερα και ε, άρα την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αποθεματικό της απόδοσης στο συμπληρώνοντας τα διευθυντικά ταμεία. Ε, για την Ιταλία, ας πούμε, έχουμε 2,5 δις. Ε, τώρα είναι δοκιμαστική λοιπόν η φάση και μετά θα μετατραπεί σε ένα μέσο, ένα tool, delivery tool, που θα βοηθήσει την εφαρμογή της, του Ταμείου Συνοχής. Δηλαδή θα είναι μια χωριστή γραμμή στον προπολογισμό. Η Επιτροπή των ε, ε, Περιφερειών συχνά έχει απόψεις που με βρίσκουν σύμφωνοι. Γιατί, Γιατί μας ανησυχεί η προσέγγιση στην ε, κεντρική διαχείριση που προκύπτει αυτό το μέτρο. Άμεση συνέπεια είναι η μετακίνηση των πόρων και των επενδύσεων από τις εδαφικέ επενδύσεις που τις διαχειριζόμασταν σε περιφερειακό επίπεδο που και τώρα μεταφέρονται σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό τόσο όσον αφορά τους φορείς, όσο αφορά και τους δικαιούχους, σε σεβασμό με την αρχή της επικουρικότητας, ε, της αλληλεγγύης και της διακυβέρνησης. Υπάρχει όμως ακόμα ένα θέμα. Άρα ενδεχόμενα περαιτέρω προβλήματα για την εφαρμογή αυτών των ε, διατάξεων πρέπει να δούμε ε, μήπως ε, τροποποιηθεί αυτό ο κανονισμό πριν από την ανάλυση τη απόδοση το 2019. Η Κομισιόν επιμένει και σήμερα στο προαιρετικό χαρακτήρα αυτή τη μετακίνηση, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει συμφωνούνται εντό εισαγωγικών με την Κομισιόν στο πλαίσιο του αποκαλούμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και άρα το σχήμα επί το οποίο βασίζεται ο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των εταίρων τη Ένωση ε, συμφωνείτε εκεί. Για τις μεταρρυθμίσεις αυτές μπορεί μέσα να συμφωνούμε. Ε, σκέφτομαι ας πούμε το είναι καταπολέμηση ε, της ε, φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής ε, και έχουμε μιλήσει και για το σύστημα της ε, πρόνοιας, ε, της υγείας που όμως οδηγεί στην επισφαλή εργασία και στην ε, επισφάλεια ε, για τον ε, εργαζόμενο κόσμο. Εμείς λέμε όχι σε όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί θα πρέπει όλα αυτά να χρηματοδοτηθούν από την πολιτική συνοχή, ακόμα και αν είναι για πρώτη φορά. Πέρα από τους πόρους λοιπόν που έχουμε βραχυπρόθεσμα, δεν συμμεριζόμαστε το νιωστό σκαμπύλι στην συνοχή. Είναι αντίθετα όλα αυτά με το στόχους ε, κοινωνικής ε, και οικονομικής συνοχής που ε, είναι γεγραμμένη στη συνθήκη. Υπογραμμίζω λοιπόν η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η αρχή της αλληλεγγύης δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τη συνθήκη και να συμφωνούμε μόνο όταν αυτό μας βολεύει. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για τη συνθήκη και όχι για το εξάμεινο παρακαλώ. Κάτι ακόμα που θέλουμε να ε, υποδείξουμε είναι ότι τα κράτη τα οποία δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν τα διαστοτικά ταμεία θα μπορούσαν για να μην χάσουν το αποθεματικό απόδοσης να ε, κάνουν εκπτώσεις και στις διαρθρωτικές αλλαγές. Και πάλι εδώ ε, ε, στην ουσία πλήττονται οι αρχές της συνοχής. Ένα ακόμα παράδειγμα, η χρήση του επόμενου μέσου για να μπορέσουμε να έχουμε μια εγγύηση για το μήνυμο εισόδημα. Για αυτή την κυβέρνηση λοιπόν για την Ιταλία είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Αν όμως κάνουμε δύο λογαριασμούς, 20 δις ε, στην ουσία τα μοιράζονται 27 κράτη-μέλη ε, και μετά οι πληθυσμοί αυτών. Είναι ένα μέσο το οποίο στην ουσία γίνεται μηδαμινό. Δεν θα ήθελα η Κομισιόν να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για μικροσκοπικές ε, παρεμβάσεις και σκέφτομαι το Wi-Fi for you που υποτίθεται θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν όλοι οι μικροί δήμοι, αλλά που τελικά κατέληξε σε μια φούσκα. Έκλεισε η προκήρυξη του διαγωνισμού ή ίσως τον Αύγουστο να ξαναγίνει και ωστόσο επρόκειτο για ψίχουλα για 27 κρατη Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι υπό την πολιτική συνοχή και τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων θα πρέπει να υπάρχει κάποια σύνδεση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο, το οποίο συνεπάγεται και σύνδεση με τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων τους ήδη έχουν κάποια project και κάποιες δράσεις που ασχολούνται ακριβώς με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να ε, υπάρχει ίση μεταχείριση. Και σύμφωνα με αυτή την ίση μεταχείριση να υπάρχουν προτεραιότητες. Ε, οι δράσεις δηλαδή και τα project που αφορούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και από την άλλη οι δράσεις που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ενέργεια, την καινοτομία, τις μεταφορές και όλα τα υπόλοιπα το αποθεματικό επιδόσεων ανταμείβει τις ε, καλές επιδόσεις. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω γιατί εισαγάγεται αυτό το νέο στοιχείο μόνο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Διότι αν ένα κρατός μέλος έχει καλές επιδόσεις, οι προτεραιότητες αυτές που ε, αφορούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, θα ε, πρέπει να είναι η αιτία ανταμοιβή αυτού του κράτους μέλους. Αντίστοιχα, αν ένα κράτος μέλος έχει καλές επιδόσεις στην ενεργειακή απόδοση, στις μεταφορές και ε, αυτό είναι προτεραιότητα στο πλαίσιο των δικών του προγράμματο μεταρρύθμισης, θα πρέπει εξίσου να ανταμείβεται για αυτές τις επιδόσεις. Επίσης, αν μας λείπει κάτι και αν βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες ελλείψεις στο αποθεματικό επιδόσεων, θα πρέπει τότε να το κάνουμε πιο ευέλικτο και να επιτεχύνουμε την ε, διαδικασία χρήσης του αποθεματικού αυτού πρέπει να ε, κοιτάξουμε όλες τις προτεραιότητες και όχι μόνο τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι η πρόταση δεν είναι καλή, διότι δεν εγγυάται ίση μεταχείριση για όλους τους τομείς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κάποιο άλλο το λόγο. Όχι, επιτρέψτε μου λοιπόν ε, κάποιες διευκρινήσεις. Καταρχάς, χρονοδιάγραμμα. Όπως ακούσατε, η Επιτροπή των Περιφερειών στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου ενέκρινε τη θέση της ε, γνωμοδότησής της. Βλέπουμε λοιπόν ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν λάθος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε και η επικάλυψη της πρότασης με την Πολιτική επιτροπή ήταν λάθος. Και υπάρχει και το θέμα της αρμόδιας Επιτροπής εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τώρα εμείς πρέπει να λάβουμε μια απόφαση, όπως και να έχει, και να την ανακοινώσουμε. Διότι ακούσαμε τη θέση της Επιτροπής των Περιφερειών, την ξέρουμε ήδη από το Φεβρουάριο, σήμερα έχουμε 20 Ιουνίου. Και δεύτερον, Πρέπει ξανά να τονίσω ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στηρίζει και εκτιμά το πρόγραμμα στήριξης των ιατρωτικών μεταρρυθμίσεων και βλέπουμε πραγματικά την αξία του προγράμματος αυτού, βλέπουμε και τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των ε, προγραμμάτων. Έχουμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας. Το ερώτημα εδώ είναι το αποθεματικό επιδόσεων. Την Δευτέρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα ψηφίσουμε την έκθεση που ε, κατάρτισε η Επιτροπή μας για το πρόγραμμα στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ε, έχουμε θετική στάση προς το παρόν στην έκθεση αυτή. Το πρόβλημα εδώ είναι, τονίζω, η χρήση του αποθαματικού επιδόσεων. και όλα τα σχόλια που ακούστηκαν από την Επιτροπή ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, σε αυτό στάθηκαν. Ε, θα δώσω τώρα το ρόλο στην Ευρωπαϊκή, ε, στο λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον κύριο Φων Μπρέσκα για ε, τις δικές του αντιδράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα... Επιτρέψτε μου να αρνηθώ την πρόταση της κυρίας Κραίλη, να αποσύρουμε την πρόταση. Θέλουμε να παραμείνει πρόταση ανοιχτή, δεν θα σας εκπλήξει αυτό άλλωστε. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι είναι προαιρετική η χρήση του μέσου. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να το χρησιμοποιήσει, κανένα κρατός μέλος. Νομίζω πως ε, όλοι θέλουμε περισσότερη ευελιξία. Και ισχύει ότι προς το παρόν τα κράτη-μέλη που ε, είναι πιο προχωρημένα στο θέμα αυτό στις συζητήσεις είναι το 6.1 και είναι η Πορτογαλία. Υπάρχουν διάφορα project ε, που δεν υλοποιούνται με τους ρυθμούς που θα έπρεπε, που έχουν χαμηλές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αποθεματικό επιδόσεων θα παρήχε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη, όταν εντοπίσουν κάποια προγράμματα που έχουν ελλειπείς επιδόσεις, να το χρησιμοποιήσουν για να διορθώσουν την κατάσταση. Εν συντομία, λοιπόν, σε λίγο καιρό μπορούν να έχουν αλλάξει ισορροπίες. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Έπειτα, ο κύριος Φανίστελ Ρόι έθιξε κάτι το οποίο είναι όντως σωστό. Έχουμε καταργήσει το αποθεματικό επιδόσεων για τις προτάσεις μας μετά το 2020. Ωστόσο, σας είπα και σήμερα το πρωί ότι θα υπάρξει ενδιάμεση αναθεώρηση το 2025. Και τότε θα έχουμε συγκεκριμένες πιστώσεις πάνω από το 6%, 14% για την ακρίβεια, πάνω από 20% λοιπόν ε, των πιστώσεων θα είναι αφιερωμένες στις αναδυόμενες ανάγκες, όπως για παράδειγμα τη μεταναστευτική κρίση που σας είπα, ακριβώς ότι κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε βάθος χρόνου και όπως ε, βλέπετε και στο, στην πρόταση κανονισμού, τις, τις συνολικές επιδόσεις, το πλαίσιο, διότι οι δείκτες εκεί δεν θα αλλάξουν. Όπως το είπε και το ηλεκτρικό συνέδριο, θα ε, εξακολουθούν να υπάρχουν, οπότε τότε θα, μπορούμε να, θα μπορούν μάλλον τα κράτη-μέλη και περιφέρειες να επιλέξουν τη δυνατότητα να αλλάξουν χρηματοδότηση και να έχουν δύο ξεχωριστές ε, πιστώσεις. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνατότητες, υπάρχει ευελιξία και θα, θα υπάρχει δυνατότητα να ανταμείβονται τα προγράμματα με υψηλές επιδόσεις. Τώρα, κύριε Βαν Μιλτενμπουργκ, πράγματι μιλάμε για καταποκοπήν ποσά. Το πώς τώρα θα καθοριστεί το ύψος των ποσών αυτών, να σας πω την αλήθεια, είναι δύσκολο αυτό να καθοριστεί από τώρα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι το αποθεματικό επιδόσεων, για παράδειγμα, στην Πολωνία είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο στο Λουξεμβούργο. Ακριβώς γιατί πιστώ στην Πολωνία είναι 80 ε, δισεκατομμύρια και στο Λουξεμβούργο πολύ λιγότερα, 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα νούμερα, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Ίσως στην πρόταση μετά το 2020 να αλλάξει αυτό. Η κατάσταση όμως τώρα έχει όπως έχει. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι δεν μπορείς να έχεις την ίδια ε, αντιμετώπιση σε όλα τα κρατημέλη διότι υπάρχουν οικονομικές διαφορές και υπάρχουν και διαφορά ταξιμεγέθους. Έπειτα είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε την αξία των μεταρρυθμίσεων. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να το κάνει δεν μπορούμε καν να αξιολογήσουμε το κόστος των μεταρρυθμίσεων, διότι πολλές φορές λέμε ότι υπάρχει κοινωνικό κόστος ε, που συνδέεται με μια μεταρρύθμιση, με αλλαγή κάποιων κοινωνικών μοντέλων κτλ. Αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον σε αυτό το πιλωτικό στάδιο, πολύ δύσκολο να καθοριστεί. Τώρα πώς σκεφτόμαστε να συνεχίσει η κατάσταση. Τα κράτη-μέλη θα κάνουν μια πρόταση ότι να αυτά θέλουμε να κάνουμε, αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αυτά χρειαζόμαστε για να τις υλοποιήσουμε και έπειτα, όπως σας είπα πριν, θα λάβει χώρο ένα διάλογος ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Θα... Ε, έχουμε προτείνει μάλιστα και έναν ε, μηχανισμό, ένα πλαίσιο αξιολόγησης ε, από ομοτήμους, όπου θα εξεταστούν τα είδη των μεταρρυθμίσεων και τα ποσά τα οποία θα ε, διατεθούν για τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Σίγουρα δεν είναι τόσο καλό, δεν είναι τέλειο, κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά σας τονίζω ότι πρόκειται για πιλωτικό πρόγραμμα και για την περίοδο μετά το 2020 θα αλλάξουν τα πράγματα. Και σίγουρα θέλετε, θα σας δώσω τώρα το λόγο για να μιλήσετε για την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων και για άλλα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω κάποια πράγματα. Τα όσα υπόθηκαν προηγουμένως ε, ισχύουν ότι Ουσιαστικά μόνο ένα κράτος μέλος, η Πορτοκαλία, θέλει να χρησιμοποιήσει το πιλωτικό. Από την άλλη, είχα ερωτήματα από μια σειρά κρατημέλη που είπαν ότι ενδεχομένω να τους ενδιέφερε να έχουν ένα πιλωτικό έργο εάν γίνει δεκτό. Και είπαν μάλιστα, ρώτησαν πόσο νωρί μπορούμε να ξεκινήσουμε το, πολιτικό, το πιλωτικό έργο. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί και από το πρόγραμμα στήριξη διαρροτικών μεταρρυθμίσεων μάθαμε ότι τα κράτη-μέλη που συμμετείχαν στην ε, προπαρασκευαστική φάση του προγράμματος υποστήριξης διευθυντικών μεταρρυθμίσεων. Ε, πιο γρήγορα πήγαιναν προς την πλήρη ενεργοποίηση του προγράμματος. Κάποια Κάποια μέλη λοιπόν ήδη τώρα ε, βλέπουν και προβλέπουν μια τέτοια δυνατότητα για το μέλλον. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό θα αφορούσε μόνο μια χώρα. Πρέπει να θίξω και ένα άλλο ζήτημα το οποίο πάντα ανακύπτει για τη συνοχή και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της ε, δημοσιονομικής κρίσης όλοι κάτι μάθαμε, ότι όταν ε, έρχεται μια τέτοια κρίση ε, μπορεί να επηρεάσει όλο τον κλάδο και όχι μόνο τον οικονομικό. Επομένω, αν δεν κάνουμε τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, θα υπάρχουν και άλλες κρίσεις στο μέλλον και θα το πληρώσουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο ζητήματα, η συνοχή ε, και οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου. Τέλος, για το ποσό που θα πρέπει ε, να δαπανάτε, όπως είπε ο Ερικ. Ναι, όντως, είναι κάτι δύσκολο. Δεν έχουμε κοστολογήσει τις μεταρρυθμίσεις, ούτε προτείνουμε κάτι τέτοιο. Το μέγεθος της οικονομικής συνεισφοράς είναι ένα οικονομικό κίνητρο, δεν μπορεί να βασίζεται στο κόστος. Σε κάποια κράτη-μέλη, σε ορισμένε περιπτώσει, ε, απαιτείται μία μεταρρύθμιση που δεν έχει μεγάλο κόστος. Απλώς δεν υπάρχει κίνητρο για την υλοποίησή τη. Οπότε εμεί θέλουμε να επικεντρωθούμε στα κίνητρα και όχι στο οικονομικό κόστος. αυτό καθ' αυτό. Και όπως είπε ο Έρικ, δεν μπορούμε να πούμε ότι η ίδια μεταρρύθμιση θα έχει το ίδιο κόστος σε κάθε κράτος μέλος. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Για κάποια κράτη-μέλη ε, αυτό έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία και σε άλλο όχι. Για την κατανομή, πράγματι θα χρησιμοποιούσαμε ε, μια αξιολόγηση ομοτήμων και εμπειρογνωμόνων για να δούμε κατά πόσο η μεταρρύθμιση αυτή θα ε, επιτύχει ε, τα παραδοτέα και ποιες είναι οι προβλεπόμενες ε, επιπτώσεις της μεταρρύθμισης. Γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε το πιλωτικό. Γιατί θα δούμε πώς όλα αυτά θα λειτουργήσουν στην πράξη πριν κατατήσουμε το ίδιο το πρόγραμμα στήριξης διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Τώρα, για τα κριτήρια αξιολόγηση βεβαίω. Ήδη ε, εμπεριέχονται στην πρόταση για το πρόγραμμα στήριξη ε, μεταρρυθμίσεων. Θα έχουμε κριτήρια για την αξιολόγηση της ε, πίστοσης υπό το πιλωτικό θα δούμε κατά πόσο πρόκειται για σημαντική μεταρρύθμιση για το σύνολο της οικονομίας, αν θα έχει λοιπόν ε, σημαντικές συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας, αν θα έχει αντίκτυπο σε ένα τμήμα της οικονομίας, αν θα είναι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, αν θα αλλάξει άρδιν ε, το μέλλον της χώρας, αν θα αυξηθεί η οικονομική αντοχή ε, της χώρας και της οικονομίας. Όλα αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να λεφτούν υπόψη λοιπόν για να καταλήξουμε σε μία εκτίμηση της πρότασης. Μιλάμε για μία μεγάλη μεταρρύθμιση, μικρή. Ε, είναι ένα κρατός μέλος που μπορεί να κάνει μόνο μία μεταρρύθμιση ή μία σειρά μεταρρυθμίσεων ε, την ίδια στιγμή για να λάβει το οικονομικό κίνητρο. Τα εξετάζουμε και τα επεξεργαζόμαστε όλα αυτά. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είμαστε σε θέση να έχουμε στοιχεία και να λαμβάνουμε ε, στοιχεία από πιλωτικά προγράμματα των κρατών μελών. Γιατί έτσι μπορούμε να δούμε πώς ε, θα βελτιωθούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Οι υπόλοιποι μιλητέ θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Ε, ναι, αισθάνθηκα την ανάγκη να παρέμβω μετά από όσα ακούστηκαν για την Πορτογαλία. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, όπως ξέρετε, ε, επηρεάζει ένα από τα μεγαλύτερα ελλείμματα που έχει η Πορτογαλία. Είναι ένα διευθυντικό πρόβλημα που έχουμε αναφέρει από το Δεκέμβριο, το είπαμε και στην Απρίλιο. Μιλήσαμε για τις ε, δεξιότητες των Πορτογάλων ε, πολιτών. Από θεωρητικής άποψης ζητάμε για το αν αυτό το κονδύλι θα πρέπει να χορηγηθεί ή όχι για τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η απάντηση θα ήταν όχι θεωρητικά. Αλλά να πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο μόνος τρόπος ε, για τις χώρες αυτές που ε, δέχτηκαν τις περικοπές στο νέο πλαίσιο είναι να έχουν μια επιπλέον βοήθεια για να κάνουν μεταρρυθμίσεις γιατί σίγουρα θα έχει μεγάλο αντίκτυπο αυτή η μεταρρύθμιση και το πιλωτικό πρόγραμμα είναι βέβαιο πως θα είναι θεμελιώδου σημασία για την Πορτογαλία και θα πρέπει να συζητήσουμε νομίζω περισσότερο αυτό το πρόβλημα γιατί εγώ φοβούμαι πολύ ότι στη δική μου μας περίπτωση της Πορτογαλίας που φαίνεται ότι είναι μοναδική περίπτωση αυτό το το πιλωτικό πρόγραμμα που αν και δεν έχει ακόμα εγκριθεί, νομίζω πως αυτές οι χώρες που χτυπήθηκαν από την κρίση δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και θα ξαναπέσουν στην κατάσταση που βρίσκονταν το 2013 και ε, πίσω. Θα πρέπει λοιπόν περισσότερο λίγο να το αναλύσουμε και να το κατανοήσουμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες που ανέφερε η Κωνσταντς είναι θέμα συνοχής και διευθυντικών ταμείων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και την ίδια την πολιτική συνοχή. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, εγώ συγγνώμη, θα, θέλω να κάνω μια σύντομη ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, γιατί μου φάνηκε πως θα έπρεπε να πάρουν το λόγο για να απαντήσουν στις δικές μου ερωτήσεις. Εσείς εκτιμάτε τα όσα λέει η Κομισιόν όσον αφορά τους λογαριασμούς, αλλά και τη λογοδοσία, ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι εγώ προτιμώ εάν συζητηθεί αυτή η πρόταση και ίσως ε, υλοποιηθεί και εγκριθεί κάποια στιγμή, προτιμώ να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου σε ένα-δύο χρόνια θα έρθετε και θα μας πείτε ότι δεν τα κάναμε καλά και ότι δεν λάβαμε υπόψη ε, συγκεκριμένα στοιχεία. Ποια είναι η γνώμη σας λοιπόν για την απάντηση που μας έδωσε η Κομισιόν. Μπορείτε κύριοι να απαντήσετε αν το επιθυμείτε ή αν προτιμάτε μπορούμε να σας στείλουμε και γραπτώ στις ερωτήσεις μας και να μας απαντήσετε σε αυτό το χρόνο. Τι προτιμάτε. Προτιμούμε την επιστολή. Μια σύντομη ωστόσο απάντηση αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται ακριβώς. Πώς ορίζονται τα ποσά. Ε, είναι, οι στόχοι πώς τίθεται, είναι μετρήσιμη; ή είναι κατά κρίση και αν είναι ε, κατά την κρίση μας, πώς μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι συμφωνούμε. Αν η Κομισιόν δεν συμφωνεί σε μια εθνική μεταρρύθμιση, αυτό σε τι οδηγεί ε, τη συζήτηση και τότε το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να έρθει και να ελέγξει τις εθνικές μεταρρυθμίσεις. Αυτού του είδους τις ερωτήσεις θα πρέπει να θέσουμε, αλλά μπορούμε να απαντήσουμε και γραπτός καλύτερα και πιο αναλυτικά. Μάλιστα, θα σας στείλουμε μια επιστολή με τις ερωτήσεις αυτές. Μάλιστα, κύριε Σπυρίδων, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν είχε σκοπό να πάρω το λόγο, αλλά νομίζω πρέπει να τονίσουμε κάποια πράγματα μετά τη συζήτηση που έγινε, που έχω την άποψη ότι έγινε σε μεγάλο βαθμό σε τεχνικό επίπεδο. Κανεί δεν είναι αντίον των μεταρρυθμίσεων. Είναι αναγκαίε. Αλλά πιστέψτε με, έχοντα κάνει μια σειρά ετών στη διοίκηση, είτε σε Δήμο, σε περιφέρειες, και σε κρατικές περιφέρειες στη χώρα μου, πιστεύω ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι μάλλον θέμα πολιτικής βούλησης της τεκάστης κυβέρνησης των κρατών μελών παρά θέμα οικονομικής ενίσχυσης. Δεν θα θέσω προβλήματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και προβλημάτων τα οποία θα φέρει μία μείωση του ποσού που είναι για, τα, για, την για, τα, για τις πολιτικές στις περιφέρειες της Ευρώπης. Θα πω όμως ότι κάτι που δεν είναι δικό μου, ο ίδιος ο κύριος Γιούνκερ το είπε, ότι η Ευρώπη περνάει μια ιδιάουσα κρίση. Κομίζω γλάφικα της Αθήνας, αν αναλύσει αυτή τη στιγμή γιατί περνάει την κρίση αυτή. Θα πω απλώς όμως ότι το μοναδικό αντίβαρο που έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα μπορούσε να έχει πολλά αντίβαρα μέχρι τώρα, το μοναδικό που έχει είναι οι πολιτικές συνοχής. Περικόπτεται λοιπόν αυτές στο επόμενο χρηματοδοτικό πολιετές πλαίσιο, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περικόπτονται γιατί διπλασιάστηκαν τα ποσά που αφορούν την έρευνα και ιδιαίτερα στην τεχνική νοημοσύνη και πολύ καλά κάναμε και τα αυξήσαμε. Περικόπτονται διότι υπάρχουν άλλε ανάγκε, όπω σχέση με το μεταναστευτικό ή με τι έκτατε ανάγκε που προκύπτουν από αυτό, την ενσωμάτωση και διάφορα άλλα παράγωγα προβλήματα. Άρα ήδη έχουμε μια μείωση των πολιτικών συνοχή. Αν εξακολουθήσει να υπάρχει άλλη μία, πιστέψτε με ότι αυτό θα είναι επικίνδυνο. Κοιτάξτε, ήμουν πρόσφατα ραπορτέρ για ένα θέμα που έχει με τις εργασιακές σχέσεις για το transportation. Ε, λοιπόν, πιστέψτε με, δεν μπορούμε να μιλάμε για ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση με τεράστιες διαφορές όταν στην Ουγγαρία ο οδηγός αμείβεται με το 1 ενδέκατο του οδηγού που αμείβεται για παράδειγμα, στο Βέλγιο. Εάν δεν κλείσει η ψαλίδα, αν δεν ενισχυθούν οι πολιτικέ συνοχή, το πρόβλημα θα είναι ουσιαστικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όλα τα άλλα θα είναι τεχνικά θέματα. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much. We are not going... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θα ξεκινήσουμε τώρα συζήτηση για την πολιτική συνοχή. Σε αυτή τη στιγμή ε, ας εστιάσουμε καλύτερα στο θέμα μας. Νομίζω αρκεί για τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους. Θα σταματήσει η συζήτηση εδώ. Έχουμε κάποιες ε, επιλογές, αρκετά πράγματα να σκεφτούμε και θα διαβουλευτούμε με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και με τους συναδέλφους για το πώς θα προχωρήσουμε. Ε, νομίζω έχουμε αρχίσει να αποκρισταλώνουμε τη θέση μας ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους πάρα πολύ. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα όμως τώρα να δώσουμε το λόγο στους διερμηνείς έτσι ώστε να επαναλάβουν άλλη μία φορά το μήνυμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και στους προσκεκλημένους μας και μετά θα περάσουμε στο τέλος της συνεδρίασης. Κυρίες και κύριοι, έχετε το λόγο.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 Thank you. This was the message uh, from the inter... Σας ευχαριστώ πολύ. To... Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε το μήνυμα των διερμηνέων και είναι σαφές πως τους στηρίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγη η συνεδρίαση και συνεχίζουμε με την συνεδρίαση των συντονιστών. Κυρίες και κύριοι, επόμενη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, Δευτέρα 25, έκτακτη συνεδρίαση και θα λάβετε ειδικό μήνυμα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ.